I think we can start. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, τελευταία συνεδρίαση για την εβδομάδα αυτή. Εχθές συνεδρίασαν οι συντονιστές. Οι αποφάσεις τους διατίθενται και αν δεν έχετε καμία διαφωνία μέχρι το 10.30 θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έχουμε το περίφημο τεστ. Αρχίζει η ψηφοφορία για να δούμε δοκιμαστικά τι γίνεται. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Όλα εντάξει. Δεν έχουμε πουθενά υπεράριθμους, όλες οι ομάδες είναι κομπλέ. Πάμε. ΕΑΣΑ. εξηγητής Μαρινέσκου. Τίτλος πρώτος, τροπολογία 1 και 245. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 1, τροπολογία 349 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 350 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 356 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 358 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 357 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 357. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ 23 κατά. 19 υπέρ 23 κατά. Παρ' όλα αυτά απορρίπτεται. 359 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 363. Εδώ έχουμε προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς με την προφορική? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν ψήφι π. Κατά αποχές εγκρίνεται. 367 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 368 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 368 έλεγχο θέλετε ορίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασα. Α, αρχίσαν οι υπεράριθμοι. Από το ΕΛΚ τώρα είναι ένας παραπάνω. Comme d'habitude. Τι έγινε, τα βρήκατε. Πέρασα. Εξοψηφία. 20-20. Ο Λιμπεράτσκι είχε πει ότι δεν έχει κάρτα. 21-20 λοιπόν εκρίνεται. Προχωρούμε. 23. Ψηφί Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. χέρι εγκρίνεται. Συμβαστική 5 είπε, Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 31 ψήφι υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. χέρι εγκρίνεται. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 391 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 392 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 396 προφορική τροπολογία διαφωνεί κανεί, Όχι. Πάμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ή 53. Έχει αποσυρθεί. 398 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 400 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 402. Όχι. Καταπίπτει. Δεν καταπίπτει. 402 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. 411 υπέρ. Όχι, ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 403 προηγουμένως και 4 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Τώρα είναι 4.11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4.12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4.16 και 17 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία 56. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές απόρριψη. 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 419 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 421 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 424 και 25 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 426 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 426 παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα πέρασε πάλι περισσεύγανες από το έλεγχο βγάλτε κάποια κάρτα So, 426. Ωραία. Πέρας. 16 υπέρ, 25 κατά απορρίπτεται. 327 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 428 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. 428 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 23 συν 1, 24 υπέρ, 16 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 4, 30 ε, υπέρ, κατά, εποχές. 4.31 προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.34 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 4.34 αρχίζει τώρα. Πέρας. 15 συν 1 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. και νέα Ψηφιπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 440 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 441 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 442 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 443 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 60 ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτό θέλει έλεγχο. Για την 60 αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. 27 27-28 υπέρ, 13 κατά. Παρακαλώ όμως να σηκώνετε και χέρι, δεν σας βλέπω. Και εκεί πίσω Μικέλε στα ορεινά. Παρακαλώ οι συζητήσει εκτός ηθούς. Ευχαριστώ. Πού ήμασταν τώρα. Τέσσερα υπέρ σου είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 466 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 467 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 470 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 471 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 472 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 473 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 473 αρχίζει. Ευχαριστώ. 20 υπέρ, 22 κατά. αποχέ καμία. Απορρίπτεται. 474 ψήφι υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. 475 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 476 υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. 477 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 478 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 479 και 480 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 483 ε, τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4, μια στιγμή. 484 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 486 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 487 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 489 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 490 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. 491 υπέρ κατά δεν τα βλέπω τα χέρια σας αποχές. Αρχίζει λοιπόν ο έλεγχος 491. Πέρας. 25 υπέρ, 15 κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. Τώρα που πάμε. 494. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ φωνές από κάτω. Λοιπόν, επαληθεύουμε το 96. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τι θα γίνει με αυτό το ΕΛΚ. Α, ήρθε ο κύριος Πίπερ, έβαλε κάρτα. Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα είστε κανονικά. Πέρα. 25 υπέρ 14 κατά εγκρίνεται. Πεντακόσια ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 503 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 504 πέ, κατά αποχές απορρίπτεται. 505 πέ, κατά αποχές έλεγχος. 505. Με η ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, 25 ε, κατά, απορρίπτεται. Και 506 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 507 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 508 υπέρ, ορίστε. θέλετε έλεγχο. Μα ήταν σαφές. Παρακαλώ, 507 αρχίζει. Πέρασε. Τι θα γίνει με το ΕΛΚ. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ κάθε φορά. Ακόμα. Ας βάλει κάποιος την κάρτα του. Oh, Τώρα είμαστε εντάξει. Πέρασε. 5 υπέρ, 35 κατά. Νομίζω ότι ήταν απολύτως απαραίτητη αυτή η επαλήθευση. Απορρίπτεται. 508 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 509 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 510 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 511 και 12 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 514 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για την 514. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. 32 υπέρ 8 κατά. Δεν φταίει ότι δεν βλέπω. Φταίει ότι δεν σηκώνει τα χέρια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, μία ώρα κάνουμε λίγο γυμναστική πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια, κάνει και καλό στην υγεία. 5-16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5-18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5-19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι σαφέστατο. 5-20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5-21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5-22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5-24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5-23 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 525 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 526 και 28, 29, 30 μαζί. Είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η 507 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 5.31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.34 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.35 υπέρ. Κατά. δεν εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 544 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 547, 47, 48, 49 και 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 551 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 556, 557, 558, 559 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60, 61, 62, 63 μαζί. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5, 64, 65 συγγνώμη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5, 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 568 κατά δεν βλέπω τι κάνετε άρχεται η ψηφοφορία επαληθεύουμε τη 568 18 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται χωρίς αποχές 569 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 569 αρχής ψηφοφορία πες 18 υπέρ, 23 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται. 567 υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω. Παρακαλώ ξανά. 5,67 υπέρ. Τώρα καλύτερα τα πάτε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5,70 υπέρ. Όχι, όχι. Ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρε. Όχι, όχι. 5, 5,70. Κατά. Αποχές απορρίψεται. 5,71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 572 υπέρ κατά αποχές φαίνεται να έχει εγκριθεί αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα είμαστε στη 572 αρχίζει η παλήθευση 16 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75, ne? Ah, Oh, falls adopted. 582. 582 κανονικά είναι η επόμενη υπέρ κατά αποχές Εφτά ψηφίσανε 582 υπέρ Κατά. Αποχές. Τώρα θέλει έλεγχο. 5.82. Αρχίζει η ψηφοφορία. geschlossen. 20 υπέρ, 22 κατά. Χωρίς αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 5,85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 586 υπέρ. Α, όχι, πέπτη. 587 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 588, 89, 90, 91, 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Μητροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 593 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 595 πάμε τώρα. Μάλιστα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 596 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 597 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 598 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 599 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 600 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 602 επέ, κατά αποχές απορρίπτεται 601 επέ, κατά αποχές απορρίπτεται 603 επέ, κατά αποχές απορρίπτεται 80 επέ, κατά αποχές εγκρίνεται 606 dafür. 606 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 605. 607 dafür. Dagegen. 607, συγγνώμη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 609 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 608 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 611 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 611 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 612 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 614 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 613 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 616 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 615 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 617 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 618 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 619 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 620 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 621 υπέρ κατά αποχές δεν ψηφίζεται. Παρακαλώ 621 ξανά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, τώρα ήταν σαφές όμως. 622 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 627 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 633 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμ... Μισό λεπτό. Ξέχασα ένα συμβιβασμό. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 643 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. 659. Ah, hm? νομίζω ότι θα πήγαινε με το. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 660 dafür. 660 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 661 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 662 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 663 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 84 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 666 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 665 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 669 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 671 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 670 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 672 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβιβαστική 21 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 66 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 678 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 679 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 680 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 681 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 682 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εξοδοντατρία, 3. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 684 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. έντεκα τώρα και 12 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές 716 7-16 Κατά. Αποχές 717 7-17 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 720 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. 726 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 24. Ψηφιπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7-35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 737 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 738 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ ορίστε 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 753 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 754 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 755 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δηλαδή εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. 756 υπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. 757 και 758 μαζί. Όχι. Καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η προηγούμενη, 139. 140 λοιπόν, υπέ, Κατά Έλεγχος. Ψηφίσουμε την 140 ηλεκτρονικά. Πέρας. 32 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 145 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 147 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 770 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 771 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 151 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 777 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 778 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 779 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 780. Ονομαστική παρακαλώ είναι αυτή. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και τελειώνει. 33 υπέρ, 8 κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. 781 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τσεκ, φωνή από κάτω. Ωραία. Αρχίζει λοιπόν ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Καλά, πλάκα μου κάνετε έτσι. Πέρασε. 17 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Εντάξει, λάθος έκανα, τι να κάνουμε. 782 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 7-83 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 784 επε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 786 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 787. Καταπίπτει. 788 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 789 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 790 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 791 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 792 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 794 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 795 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 801 υπέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 802 υπέ. κατά αποχές απορρίπτεται. Οι τροπολογίες 803 και 804 μαζί υπέ. κατά αποχές εγκρίνονται. 807 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 808 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 809 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 810 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές 811 8-11 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 812 ειπε κατά αποχές εγκρίνεται. 813 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 ειπε κατά αποχές εγκρίνεται. 182 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 814 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 815 υπέρ. Τσεκ για την 814. Ορίστε, αρχίζει τώρα. Πέρας. 30 υπέρ, 13 κατά, χωρίς αποχές εγκρίνεται. 8.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές 8 16 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 λέει ο πρόεδρος, ε, δηλαδή 185, ευχαριστώ πολύ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 819 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 820 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 821 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 822 και 823 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 824 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 825 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 και 826 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. «188-827 μαζί, αρχίζει η ψηφοφορία». Ist geschlossen. 20 dafür. 20 υπέρ, 21 κατά και μία αποχή απορρίπτεται. 188 Αυτό ήταν 187 και 826. Τώρα πάμε 188 και 827 υπέρ κατά. Και αυτό θέλει έλεγχο. Δεν ψηφίζεται. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 21 υπέρ 19 κατά. Μια αποχή εγκρίνεται. 828 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 829 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 832 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 833 83επε κατά αποχές απορρίπτεται. 834 επέ κατά αποχές απορρίπτεται. 835 επέ κατά αποχές εγκρίνεται. 836 επέ κατά αποχές εγκρίνεται. 837 υπέρ κατά, αποχές, απορρίψετε. 8.38 Είπε κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8.38, έλεγχο θέλετε παρακαλώ. Πέρας. 23 υπέρ, 20 κατά, χωρίς αποχές εγκρίνεται. 839 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οκτώ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 845 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 846 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «854 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω χέρια να σηκώνονται ξανά 854 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 857 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 858 υπέρ όχι όχι καταπίπτει αυτή και η επόμενη. 35 λοιπόν συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 862 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 865 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 866 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 867 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 37 υπέρ. Ονομαστική, συγγνώμη. Αρχίζει τώρα λοιπόν, που είναι ονομαστική. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. 37 υπέρ, 5 κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. Κομπρομίς 38. Dafür. 30 συμβαστική, 38 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8,96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «898 ειπε κατά, εποχές εγκρίνεται». «899 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 900 υπέρ, όχι. Ναι, 900 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψεται. Α, όχι, καταπίπτει 900. Ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρος, επειδή κρίναμε την 899. Ωραία. Άρα τώρα πού πρέπει να πάμε. Όχι, σωστό ήτανε. Λοιπόν, πάλι, πάμε πάλι. Ψηφίζουμε την 900 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 901 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 904 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 905 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται 906 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται 908 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 907 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται 909 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 910 και 11 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 912 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 913 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 914 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική 915. διαφωνεί κανεί με την προφορική, όχι. Τι ψηφίζουμε λοιπόν, έτσι, με την προφορικη είπε υπέρ, κατά, αποχές, 916 9-16 υπέρ, κατά, αποχές, 917 9-17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 920 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Ε, ελέγχουμε την 920 Αρχίζει της προφορίας. 14 υπέρ, 26 κατά η μία αποχή. Απορρίπτεται. 921 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 922 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 923 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 924 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 924 έλεγχος παρακαλώ αρχίζει ψηφοφορία στην 924 ist geschlossen. 9 dafür, 32 dagegen. 9 υπέρ 32 κατά, χωρίς αποχές, απορρίπτεται. Και αυτή η πολύ σημαντική επαλήθευση. Ε, 925 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 41 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 926 υπέρ όχι 29 συγγνώμη, κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι 229. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 930 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9.33 ε, και 9.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9.35 και 36 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 208 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δυτικό 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9.43 και 44 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι έγινε. Hm? Πού είμαστε τώρα στη 16-17. bis... Α, μπορούμε να τα ψηφίσουμε unblock τώρα όλα αυτά. Συμφωνείτε του κυρίου Μαρινέσκου από 2.17 μέχρι 9.49 όλες μαζί. Ο μου που λένε. Α, μέχρι το 2.25 τότε. Ωραία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται όλες αυτές. 9.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9.49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9.50 και 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9.56 και 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «972 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 231 είμαστε τώρα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 973 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 977 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 978 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 932 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 48 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 933 και 983 μαζί είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 984 ε, είπε. κατά έλεγχος. 984 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. 9,85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9,86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9,87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9,88 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 989 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 990 και 991 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 992 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 993 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 και 95 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. 96 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Τι να κάνουμε, δεν σηκώνεται χέρια. 998 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασα. 17 υπέρ 24 κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 1000 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 1002 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1005 και 1006 μαζί υπέρ. 1002 δεν την εγκρίναμε. Α, δεν την ψηφίσαμε. Τι γίνεται τώρα. 1008, 1009, 1010 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1013 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1014 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ γιατί 1014 αρχίζει τώρα Πέρας. 17 υπέρ 24 ε, κατά απορρίπτεται. 1015 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χίλια σαράντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1043 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1044 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1045 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1046 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 463 υπέρ κατά κατά αποχές δεν βλέπω τι κάνετε 463 ηλεκτρονική υπολήθευση αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας. 6 υπέρ 36 κατά. 37. Χωρίς αποχές απορρίπτεται. Σας παρακαλώ, σηκώντε τα χέρια σας. Δεν είχα δει τίποτα προηγουμένως πριν. 462 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, όχι, όχι. Ως προσθήκη λέει. Μόνο προσθήκη είναι. Την ξαναψηφίζουμε υπέρ. 462 κατά αποχές εγκρίνεται. 485 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται. Συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1049 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 1050 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1051 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1052 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1053 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1054 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, έλεγχο θέλετε για τη 1054. Παρακαλώ, αρχίζει η παλήθευση. Πέρας. 18 υπέρ, 25 κατά. Χωρίς αποχές απορρίπτεται. 1055 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 237 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1056 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1059 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 55 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 1061 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 1062 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 1063 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 1064 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 1065 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1066 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1067 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι τοπολογίες 572 και 588 έχουν απορριφθεί. Ψηφίζουμε τις άλλες δύο υπέρ, 68 και 69, 1068 και 1069. Όχι, αφού δεν λέει καταπίπτουν, λέει ο κ. Βάντεμ αν έχουν απορριφθεί άλλε δύο. Α, μάλιστα. Άρα καταπίπτουν και οι δύο αυτές γιατί έχουν ε, απορριφθεί οι δύο προηγούμενες. Άρα πάμε 1070 και 1071 τώρα. Υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτουν. 1072 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1073 τσεκ 1072 αρχίζει η επαλήθευση πέρασε 35 υπέρ 9 κατά εντάξει εγκρίνεται λοιπόν 1073 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1074 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1075 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1076 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1077 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1078 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1079 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1080 και 81 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1082 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 56 υπέρ, κατά, ο, ξανά. Συμβαστική 56 υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1088 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1092 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1093 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1097 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1098 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1100 dafür 1100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1112 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 246. 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 60 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 3.42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 64 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 280 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τσεκ 280 ορίστε παρακαλώ αρχίζει. Πέρας. 20 υπέρ 23 ε, κατά απορρίπτεται. Λοιπόν, συμβαστική 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 294 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 303 είπε κατά αποχές απορρίπτεται 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 313 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 317 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 322 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Αρχίζει τώρα για την 322. Πέρας. 20 υπέρ, 23 κατά χωρίς αποχές, απορρίπτεται. 323 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 324 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία τριάντα υπέρ κατά φόλους φωνές. Μα δεν εγκρίθηκε 280, δεν καταπίπτει καθόλου. Εντάξει. 331 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 331. Πέρας. 20 υπέρ, 22 κατά, χωρίς αποχές, απορρίπτεται. 3, 32 και 333 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 334 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.36 υπέρ καλά κατά αποχές έλεγχος 3.36 αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε. 17 υπέρ 25 κατά μία αποχή απορρίπτεται. 3.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 340 υπέρ κατά ξανά κατά εγκρίνεται αποχές εντάξει ε, η 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 341 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.43 33π ναι. Τα ίδια με πριν ισχύουν. 3.43 είπε Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 3.43. Ελέγχουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 23 κατά χωρίς αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, ακολουθεί η τελική ψηφοφορία ονομαστικά, καταρχήν. Ένας. 31 υπέρ, ένας κα... 11 κατά, μία αποχή και εγκρίνεται. 11 31 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή. die Τώρα θα ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα, αρχίζει η ψηφοφορία. και τελειώνει με την ίδια πλειοψηφία, 31, 11 και μία αποχή, 32 συγγνώμη, ναι. Και τώρα θα ψηφίσουμε την διαπραγματευτική εντολή. Εδώ χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 32 υπέρ, 10 κατά, 2 εποχές. Ωραία. Δίδεται και η εντολή. Και τελειώσαμε αυτή την έκθεση. Συγχαρητήρια. Gratuliere Συγχαρητήρια στον εισηγητή, κύριε Μαρινέσκο. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και τη γραμματεία Τραν και ιδιαίτερα τον Σφεν Ότ, ο οποίος είναι και άρρωστος κανονικά και έχει προετοιμάσει ε, την ψηφοφορία αυτή με αυτό το τέλειο τρόπο, τρομερή ευσυνειδησία. So we will continue. Please leave the room or sit down, please. Αν θέλετε να αποχωρήσετε παρακαλώ ησύχως. Now we continue. Please sit down or leave the room. Παρακαλώ, ε, συνεχίζουμε. Είτε θα καθίσετε, είτε θα βγείτε από την αίθουσα. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τώρα ε, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναύση πλοία. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκεζίνε Μάισνερ και ψηφίζουμε την τροπολογία 117 για αρχή. Ψήφι υπέρ αποχές απορρίπτεται. Sit down. In any case, be... Παρακαλώ ησυχία. Και άμα θέλετε να φύγετε, φύγετε. Και άμα θέλετε να καθίσετε, καθίστε. Εντάξει, πιάνει και όλα, είδατε. 119, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 119. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. 12 υπέρ, 28 κατά. Με μία αποχή. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. 118 μάλλον. 119 ήταν αυτή. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν κρίνεται. Θέλετε έλεγχο για την 118. Αρχίζει λοιπόν ο έλεγχος. Ελεκτρονική παλιδεύση. Πέρασε. 15 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Αρχίζει η παλήθευση. Πέρασε. 29 υπέρ, 11 κατά. 29 συγγνώμη. Και μία εποχή. Εγκρίνεται. 130 και 131 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετροπολογία, ναι, υπέρ. Εντάξει, τώρα ήταν μεγάλη πλειοψηφία. Τι θέλετε. 9 ε, υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. Έμπλου 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εμπλήκωση υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 135 και 136 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 21, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Παρακαλώ. Αρχίζει τώρα. Ψηφίζουμε την 21 της Επιτροπής Αποσχόλησης. Πέρασε. 13 υπέρ 27 κατά. Χωρίς αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Έμπλου 22 υπέρ κατά. Αποχές έλεγχος. 22 της Επιτροπής Απασχόλησης αρχίζει τώρα. 15 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. 138, 140 και 41 μαζί, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142, 143, 144 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά. Δεν τα βλέπω. Ε, ελέγχουμε λοιπόν για τη 12. Πέρας. 24 υπέρ, 16 κατά, ε, χωρίς αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 8, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά, αποχές, έλεγχος. Ελέγχουμε τη συμβαστική παρελθόν 2, αρχής ψηφοφορία και τελειώνει. 22 υπέρ, 16 κατά, με δύο αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές Έλεγχος 147 αρχίζει τώρα η επαλήθευση. Πέρασε. 24 υπέρ, 13 κατά χωρίς αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 ε, της απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλου 25 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 25 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 26 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 27 είπε, κατά αποχές έλεγχος. 27 της Επιτροπής Απασχόλησης αρχίζει. Πέρας. 14 υπέρ, 27 κατά, χωρίς αποχές απορρίπτεται. Τοπολογία 27, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 11 κατά πίπτη, έμπλη 28 υπέρ, κατά αποχές απόρριπτου. 169 και 170 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Έμπλε 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 37. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 40. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 εμπλυπέ κατά αποχές έλεγχος. Τη 40 της Επιτροπής Απασχόλησης ψηφίζουμε τώρα. Λέξεις 16 υπέρ, 25 κατά, δύο αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 41 υπέρ, κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιούρι 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 194 είπε. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 46 και Γιώργη 18 είπε. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 47 και Γιώργη 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιώρη 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 214 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 215 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 είπε. Κατά. Αποχές έλεγχος. 54 ελέγχουμε παρακαλώ. Αρχίζει τώρα ηλεκτρονική απολύθευση. Πέρασε. 10 υπέρ, 29 κατά, 3 αποχές. Καταλαβαίνω ότι έχετε κουραστεί λίγο να σηκώνετε κανένα δάχτυλο. Γιούρι 23, υπέρ. Κατά. Πάλι δεν βλέπω τι κάνετε. Ξανά, 23 υπέρ της Γιούρι κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Γιούρι 23. Αρχίζει τώρα η επαλήθευση. Πέρα. 15 υπέρ, 16 δηλαδή, 25 κατά. Θαυμάσια. Α, πραγματικά δεν φαινόταν έτσι που δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Απερίφθη. Ωραία. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αυτά είναι σαφή πράγματα. Τώρα, έμπλη 43. Ε, Είμαστε στα παραρτήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 18 υπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέ, κατά αποχές Νομίζω θέλει έλεγχο τώρα αυτή. η 251 αρχίζει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 22, 23 υπέρ, 18 κατά και 2 εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 252 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Η τροπολογία 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 2 υπέρ κατά έλεγχος. Έμπλ 2 την επαληθεύουμε παρακαλώ αρχίζει η προφορία. 19 υπέρ 22 κατά δύο αποχές απορρίπτεται. Χωριστή ψηφοφορία στην 75. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλη 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, ξανά υπέ κατά, αποχε έλεγχος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία και τελειώνει. 23 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Η τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ορίστε. 85 υπέ. Κατά. Αποχές. Και αυτό θέλει έλεγχο. Για την 85 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. 19 υπέρ 21 κατά μία αποχή απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Γιούρι 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άμπλ 5 υπέρ κατά αποχές αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε. Αρχίζει ο έλεγχος ηλεκτρονικά. Πέρας. 14 υπέρ, 26 κατά, με δύο εποχές απορρίπτεται. Από ψηφίπε, ψηφί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άμπλη 6 υπέρ, κατά. Και πάλι δεν βλέπω τι γίνεται και δεν τσεκάρω. Έμπλο 6, αρχίζει η ψηφοφορία. 14 υπέρ, 26 κατά. 15 δηλαδή υπέρ, 26 κατά και δύο εποχές Απορρίψετε. Η τροπολογία είναι 90 υπέρ. Κατά, εποχές απορρίψετε. Η τροπολογία είναι ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εμπλεπτά υπέ. υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Εμπλοκτό υπέ. κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ορίστε. 92 να την ελέγξουμε, παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. 16 υπέρ, 26 κατά, απορρίψετε. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμπλε 9 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Έμπλε 9 αρχίζει η ψηφοφορία η οποία τελειώνει κιόλα. 15 υπέρ, 26 κατά, δύο εποχέ απορρίπτεται. Έμπλ 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά. Δεν σας βλέπω τα χέρια σας. Αρχίζει λοιπόν η επαλήθευση. Ist geschlossen. Πέρας. 16 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται. Γιούρι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άμπλη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιώρη 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην τελική ψηφοφορία που είναι και με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Πέρας. 35 υπέρ, 4 ε, κατά, 2 εποχές. Θα πρέπει να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα μετά. Και πάλι με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Πέρας. 35, 36 υπέρ 4 κατά 2 εποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στις διαπραγματεύσεις και χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για την εντολή. Αρχίζει τώρα. Η ψηφοφορία. Πέρας. 35 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια Γκεζίνε Μάισνερ. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Jahresbericht über die Wettbewerb. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την αιτήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Bericht von Econ und είναι ε, ε, η συγκήτρια Τζάκλιν Φώστερ, γνωμοδότηση είναι αυτό. Συμβιβασμός παριθμών 1, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά έλεγχος για την τροπολογία υπαριθμών 6 αρχίζει τώρα. Ist geschlossen. 19 dafür. 19 υπέρ, 19 κατά ισοψηφία και μία αποχή απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Την τροπολογία 11 αρχίζει. Τέλος. 17 υπέρ 20 κατά 2 αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 2 ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25, καταπίπτει, όχι, όχι, υπέρ. Ναι, ναι, φόρος καθόλου, γιατί δεν εγκρίθηκε 24. 25 λοιπόν ψηφίσμα υπέρ. Κατά 25, επαναλαμβάνω, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τσεκ, ωραία, το ελέγχουμε. Επαληθεύουμε λοιπόν την 25. Πέρας. 20 18 κατά. Χωρίς αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχο θέλετε για την 32 ορίστε αρχίζει Πέρασε. 16 υπέρ, 23 κατά απορρίπτεται. Μάλιστα. 33 υπέρ, κατά. Και αυτό θέλει έλεγχο όμως τώρα. Αρχίζει ο έλεγχος για την 33. Πέρας. 16 υπέρ, 21 κατά, δύο εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία στην 41. Τμήμα πρώτον, υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, τσεκ. Το δεύτερο τμήμα το ελέγχουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία στη 41 τροπολογία. Πέρασε. 17 υπέρ, 22 κατά. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 5 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό το ελέγχουμε γιατί 49 αρχίζει. Πέρασε. 19 υπέρ, 19 κατά και μία εποχή απορρίπτεται. Η τροπολογία 50 ψήφι πε Κατά. Αποχές. Και αυτό θέλει έλεγχο. 50 αρχίζει τώρα. Πέρασε. 20 υπέρ, 19 κατά χωρίς αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Η 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές δεν σηκώνεται χέρια. 52 υπέρ. Α, ορίστε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Όχι, καταπίπτει αυτή. Όχι, δεν καταπίπτει. Είπε 53 κατά. Αποχές απορρίψετε. 54 είπε Κατά. Αποχές. Τσεκ. Το 54 λοιπόν ελέγχουμε παρακαλώ. Αρχίζει. Πέρασε. 16 υπέρ, 20 κατά. Οι τρει αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Η τροπολογία 60 υπέρ, κατά, Ελέγχω παρακαλώ. Η τροπολογία 60. Αρχίζει τώρα. 15 υπέρ, 20 κατά, 4 αποχές η τροπολογία 63. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε Η τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό το ελέγχουμε. 62 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ 17 κατά. Α, 19 υπέρ 17 κατά και μία εποχή. Εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά υπέρ μάλλον ξανά κατά έλεγχος. το 75 αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασα. 16-17. Μπορεί ο Φιλιμπεράτης και τι ψηφίζει. 16 υπέρ, 19 κατά. Και τρεις αποχές. Απορρίπτω. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, απόχέ. έλεγχουμε. Την 79 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. 19 υπέρ 19 κατά ισοψηφία, μία αποχή, καμία αποχή μάλλον, απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 82 υπέρ, κατά αποχές συγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, έλεγχος. 83 λοιπόν, αρχίζει τώρα. 17 υπέρ, 20 κατά, 2 αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Πέρασε. 28, 29 είπε, 10 αποχε... ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Φώστερ. Hm ich Επόμενη ψηφοφορία της έκθεσης σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕΠ. Έκθεση Λιμπεράτσκι. Νομοδότηση δικιά μας είναι. Συμβαστική ένα ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ γιατί την 56 αρχίζει τώρα η παλήθευση. Περάσει. 15 υπέρ 23 κατά. Ορίστε. Δεν δουλεύει το μηχάνημά σας, κύριε σας όλοι. Χωρίς αποχές απορρίπτεται. Η τροπολόγια 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 καταπίπτει. Πάμε στην 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά έλεγχος. Την 59 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. 20 18 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι δεν είναι. Με υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά από η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Την ελέγχουμε όμως ηλεκτρονικά, αρχίζει τώρα. Πέρας. 7 υπέρ, 26 κατά. Ευχαριστώ για τον έλεγχο, Βιμ. Αλλά καμιά φορά φαίνονται τελείως ανάποδα τα πράγματα. Είναι τρελά. Μα ποτέ δεν, δεν μέσα, λέει ο Βαντεγκάπ. Όχι και ποτέ. 13 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. ist geschlossen. 33 υπέρ, όχι 34 υπέρ με τον εισηγητή, 3 κατά δύο εποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, Μπόγους Λιμπεράτσκι. Mhm. Τώρα έχουμε τη ρομποτική του Γκέορκ Μάγερ. κανόνε αστικού δικαίου σχετικά με τη ρομποτική. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την συμβαστική υπέρθμον 1 αρχίζει τώρα. Ist 21 υπέρ 7 κατά χωρίς αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την συμβαστική 3. Αρχίζει τώρα. Μα έλεγχο κάνω. Αφού θες έλεγχο, τι γελάτε. Πέρας. 21 υπέρ 7 κατά χωρίς αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ. Dagegen. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά Έλεγχος. 19. Αρχίζει τώρα. 21 υπέρ, 7 κατά, χωρίς αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 32 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 είπε, Όχι. Η συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. χέρι εγκρίνεται. Η 44 είπε, Κατά. χέρι εγκρίνεται. Συμβαστική 6 είπε, Κατά. χέρι εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. χέρι εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Από ποια συγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Τι τσεκ, τι να τσεκάρω. Την 75, ωραία. Αρχίζει η προφορία. Πέρας. 7 υπέρ, 21 κατά, χωρίς αποθήκες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρα κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρα κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τι τσεκ, το 4 θέλετε να τσεκάρουμε. Αρχίζει λοιπόν τώρα ο έλεγχος. Πέρας. 13 υπέρ, 15 κατά. Χωρίς αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3 ελέγχεται και Επαληθεύεται ηλεκτρονικός. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, 1 κατά, χωρίς αποχές. Καλά που το τσεκάραμε, έτσι. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρας. 22 υπέρ, 5 κατά, χωρίς αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, δεν μπορώ να δώσω στον εισηγητή διότι απουσιάζει. Τελευταία ψηφοφορία. Ε, είναι η τέταρτη δέσμη. Όχι, δεν είναι τα σιδηροδρομικά, όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εφαρμογή τη αρχή τη μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Προηγουμένω τα λέγαμε κύριε σας όλοι για τα συνδρομικά, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Εφαρμογή τη αρχή τη μεταχείρισης και τα λοιπά στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε και την παροχή αυτών. Η Συνογέννη Νίλσον. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απο, εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές. Ξανά. 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 15 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 16 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 17 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 19 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Πέρας. 32 υπέρ, 4 κατά μία αποχή εγκρίθηκε 33 με τον κύριο Λιμπεράτσκι. Ε, συγχαρητήρια κύριε Νίλσον. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει μία ώρα. Παρακαλώ, ή καθίστε ή φύγετε από την αίθουσα. silent. Και ησυχία πάνω απ' όλα. Πάμε στο επόμενο θέμα στη μέσα διάταξη. Τώρα είναι το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Δεύτερη ανάγνωση για τη διάνοιξη της αγοράς, διακυβέρνηση συνδρομικής υποδομής και συνδροματικών επιβατών. Ο Βίμ Κάμπ, ο Σασόλη και η κυρία Κίλωνεν είναι εισηγητές. Θα δώσω πρώτο το λόγο στο Βίμ Κάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που επέζησα σε αυτές τις τεράστιες πληροφορίες έτσι τόσο μακροσκελής. Πάρα πολλές πληροφορίες τώρα τόσες ώρες ψηφίζουμε εδώ πέρα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τμήμα PSO του τετάρτου πακέτου ιδέσμης και ιδιαίτερα το πολιτικό για τη διαχείριση, πρέπει να σας πω ότι έκανα πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις και στην Ολλανδική Προεδρία στις 19 Απριλίου ενεστώτος έτους συμφωνήσαμε. Η συμφωνία αυτή είναι καλή. Τρία ήταν τα σημεία που μας ενδίεφεραν, ήταν το άνοιγμα της αγοράς πρώτα απ' όλα. Ορίζει λοιπόν το PSO ότι καταρχήν όλα τα σιδηροδρομικά ταξίδια και οι διαδρομές και τα δρομολόγια θα πρέπει να προκυρήσονται ε, σε διαγωνισμό, ε, αλλά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις από τους ε, πληστηριασμούς αυτούς έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται αναθέσεις άμεσες χωρίς διαγωνισμό. Αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος της αγοράς, κυρίως κάποιες ιδιαιτερότητες περιφερειακές και γεωγραφικές. Αλλά στην άμεση ανάθεση οι εθνικοί επόπτες οι αρχές δηλαδή, θα πρέπει να εξετάζουν κατά πόσο γίνονται σωστά και σύνομα όλα αυτά, ακόμα και στις άμεθες αναθέσεις. Και μήπως έπρεπε να γίνει διαγωνισμός και τους δόθηκε χωρίς διαγωνισμό. Αυτό ήταν το πρώτο που κυριάρχησε στις διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα τροχαίου υλικού. Δηλαδή κάποιος κερδίζει το διαγωνισμό. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει το διαγωνισμό, αλλά αν δεν έχει τρένα, τι να την κάνεις αυτή που κέρδισε. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν αν υπάρχει αγορά leasing για εκείνο που κέρδισε το διαγωνισμό. Γιατί σας είπα, ωραία, κατεβαίνεις υποψήφιος, κερδίζει ένα διαγωνισμό, δεν έχει τρένα να βάλεις τη διαδρομή στο δρομολόγιο που κέρδισες και θα το κάνεις τι. Το τρίτο σημαντικό, ε, πρόεδρε, ήταν τα κοινωνικά στοιχεία και οι κοινωνικέ πτυχές των δημοσίων διαγωνισμών και του κανονισμού PSO. Το Συμβούλιο ήταν τρομερά άκαμπτο σε σχέση με αυτό αλλά εμείς καταφέραμε στην εθνική νομοθεσία ε, να ε, ισχύουν όσα ισχύουν για τους εργαζομένους και αυτό να κυριαρχεί. Και όταν κάποιος αναλαμβάνει κάποιες συμβάσεις προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το PSO που είναι υποχρεώσεις δημοσίου τομέα, ε, κοινοφελούς υπηρεσίες, public service obligations, για τις άμεσες αναθέσεις, για την ε, ε, ύπαρξη τροχαίου υλικού, σειρμών δηλαδή, και για τις κοινωνικές ψυχές και την προστασία όταν κάποιος κερδίζει τη σύμβαση. Αυτά. Καλή είναι η συμφωνία, βέβαια δεν τα περάσαμε όλα, αλλά επαρκεί έτσι ώστε να κάνουμε και το επόμενο βήμα για να ανοίξει η αγορά στην Ευρώπη για τα τρένα. Και να μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ όμως να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε τρομερή πίεση χρονική. Κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχω ξαναπεί. Ε, το να το να συνεργάζεται κανεί με τον κύριο Φάντεν Κάμπ είναι πραγματική ευχαρίστηση, παρόλο που υπάρχουν κάποιε αποκλήσει στι απόψει. Η δική μου η αποτίμηση του θέματο είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Ε, διότι υπάρχουν κάποιοι βασικοί τομεί που θα πρέπει να καλύψουμε, όμω υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσβαση, επίση κοινωνικέ πτυχέ σε σχέση με την εθνική νομοθεσία Δική μας πρόθεση είναι να προβλέψουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία για τους πολίτες και να μην αναφερθούμε στην ε, νομοθεσία των επιμέρους χωρών. Ε, τώρα ε, για, το σχέδιο αυτό, για αυτή την έννοια, το Public Service Obligation της υποχρεώσεως κοινοφελών υπηρεσιών, ε, Θέλουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη για τις υδροδρομικές μεταφορές ή θα είναι πολύ συγκεκριμένη η διαδικασία όπου θα προβλέπουμε τον τάδε αριθμό ε, αμαξοστοιχειών για τον τάδε αριθμό επιβατών και θα κανονίζουν ξεχωριστά η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο λόγω χάρη θα κάνουν. Ε, εάν κοιτάξετε το τελικό αποτέλεσμα των συζητήσεων στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, τι βλέπετε, η τελική πρόταση στο σημείο 1 αναφέρει άμεση υποχρέωση θέση του Συμβουλίου για την μεταβατική περίοδο. Έχει βρεθεί ένα μια συμβαστική λύση. Για τα κοινωνικά θέματα, θέση του Συμβουλίου, ε, ρήτρα αμοιβαιότητα, μικρομεσαίε επιχειρήσει, προγράμματα μεταφορά θέση του Συμβουλίου, βιομηχανικό απόρριτο. Αυτή είναι η κοινή θέση. Και μετά υπάρχει μια σειρά από ειδικέ προποθέσει, όπου εμεί ω Κοινοβούλιο έχουμε ακολουθήσει τελείω αμυντική στάση. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο επί το οποίο το Κοινοβούλιο να μπορεί να πει ότι στι διαπραγματεύσει ελήφθη υπόψη η άποψή του. Κατά την άποψή μου αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Ευχαριστούμε κύριο Στελίτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Οι δικές μου προσδοκίες ήταν κάπως διαφορετικές και πιστεύω ότι καμιά φορά αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε όπως θα θέλαμε. Η διάκριση που γίνεται μεταξύ των όσων λέγονται και όσων τελικά ε, κάνουμε πράξη στο Συμβούλιο, πόρο απέχουν ε, μεταξύ τους. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι για τα κοινωνικά πρότυπα διαφέρω κάπως τις απόψεις μου από τον καλό φίλο κύριο Λιμπεράτσκε και θα έλεγα πως μόνο τόσο μπορούσαμε να καταφέρουμε όχι μόνο μεταξύ ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν ε, κοινωνικές επιπτώσεις είτε για αυτού που κερδίζουν μια ανάθεση είτε για αυτού που χάνουν ένα συμβόλαιο. Και το γεγονός πως μιλάμε για εθνικά πρότυπα και έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά τη γνώμη μου με δυσκολία θα στηρίξουμε, γιατί βεβαίως οι προσδοκίες μας αρχικά ήταν υψηλότερες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντέλη και μετά η κυρία Νοτζή. Κυρία Νότζου, θα ήθελα να σχολιάσω και τις τρεις εκθέσεις παράλληλα. Να το κάνω τώρα ή αφού ακούσουμε και την παρουσίαση για την τελευταία έκθεση. Έτσι ώστε να συντομεύσω. Μετά, στο τέλος. Ωραία, λοιπόν θα τα πω στο τέλος. Κύριε Σασόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτέλους και εγώ μπορώ να παρουσιάσω το τελικό σχέδιο μετά από τη δεύτερη ανάγνωση και θα ξεκινήσω την ε, ομιλία μου ευχαριστώντας όλους και για μένα είναι μεγάλη χαρά να μπορώ να συνεργαστώ με τον Βιν Φαντερκάμπ αλλά και όλους τους συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με αυτή τη δέσμη μέτρων για τους ίδριοδρόμους. Την κυρία Κιλόνεν, το φίλο μου, τον κύριο Λιπεράτσκι. Ευτυχώς έχουμε συνεργάτες και συναδέλφους στην Επιτροπή με μακρά πείρα που μας ε, συνόδευσαν σε όλη αυτή την μακρά πορεία. Ξέρετε ότι ο Τιμαρής διάλογος κράτησε πολύ καιρό, ήταν ιδιαίτερα περίπλοκος αλλά πρέπει να ευχαριστήσω και την Ολλανδική Προεδρία, διότι καταφέραμε να βγάλουμε την κατάσταση από το τέλμα στο οποίο βρισκόταν και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που θεωρούμε θετικό από τη δική μα την οπτική γωνία ε, για, την, ε, για τον κλάδο των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Είναι ένα βήμα πρόοδου ώστε να καλύψει την ε, διαφορά του με τον τομέα των αερομεταφορών. Δεν είναι απλό όπως θα ξέρετε, διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πολλές εξαιρέσεις οι οποίες επισημάνθηκαν ως ανάγκη από πολλές κυβερνήσεις κρατομελών μελών και θεώρησα παρατητό να αναγνωριστεί λόγω της ιδιαιτερότητας και της ομογένεια του σιδηροδρομικού κλάδου, ε, το σύνολο αυτό των εξαιρέσεων. Μπορώ να πω ότι σήμερα, χάρη σε αυτή τη δέσμη μέτρων, θα υπάρχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην Ευρώπη και ότι δικέ μα επιχειρήσει και εταιρείε θα έχουν όλε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν τι υπηρεσίε του. Θα υπάρξει σαφώ βελτίωση αυτών των υπηρεσιών. Μείωση των τιμών για τους ταξιδιώτες, τους επιβάτε και περισσότερες επιλογές. Επιλογές τη στιγμή της κράτησης ε, εισιτηρίων και ταξιδιών. Να θυμίσω σε όλους ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου εδώ ήταν ε, καθοριστική σημασία για την επίταξη συμφωνίας στο Συμβούλιο. Συμφωνίας που έπρεπε να γίνει με κριτήρια την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των φορέων του δικτύου καθώς και το άνοιγμα της πριν από το άνοιγμα τη αγορά των σιδηροδρόμων. Ε, το Κοινοβούλιο λοιπόν επιδίωξε του εξή στόχους. Πρώτον, προβλέφθηκαν μέτρα διαφύλαξη προκειμένου να βεβαιωθούμε για την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των διαχειριστών των υποδομών, ενισχύοντα τι διατάξει που έχουν να κάνουν με τις διπλές ε, εντολές τις βασικές αρμοδιότητες, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τον προγραμματισμό της συντήρησης την ε, εξωτερήκευση, εξωτερική ανάθεση δηλαδή, και την ε, ε, κατανομή των λειτουργιών του κεντρικού διαχειριστή των υποδομών. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν ένα εθνικό πλαίσιο κανόνων για την αξιολόγηση των συγκρούσεων συμφερόντων, εντός του οποίου οι ρυθμιστικοί οργανισμοί, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη ε, το προσωπικό συμφέρον που μπορεί να έχει οικονομικό, ε, χρηματοοικονομικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα και θα μπορούσε εσφαλμένα ε, και κακώς να φύξει την αμεροληψία του διαχειριστή. Τρίτον, έχουν ε, συνταχθεί ειδικέ ε, διατάξεις για να διευθετηθούν οι κανόνες πρόσβασης ε, των επιβατών των αμαξοστοιχειών υψηλής ταχύτητας στο υλικό του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο δίκτυο υψηλής ταχύτητας ακριβώς και να προωθηθεί ανταγωνιστικότητα προς όφελος αυτών των ιδίων των επιβατών. Τέταρτον, κοινωνικές πτυχές. Ένα θέμα πολύ θερμό και πολύ κέριο. Ε, για μένα επίσης πολύ σημαντικό μια σιδηροδρομική επιχείρηση που θα απαιτήσει μία έκδοση τη οποία ή της οποίας η υπευθυνη ε, δεν θα πρέπει να καταδικαστεί σε ποινικέ κυρώσεις στην περίπτωση που ε, προβλέψει ε, εξαιρέσεις από συλλογικέ συμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δεσμευτικές. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να ε, προβλέψει κανόνες προστασίας για το προσωπικό του σιδηροδρομικού δικτύου. Επίσης, πέμπτο σημείο, ε, ειδικέ μορφές συνεργασίας των διαχειριστών του δικτύου με, όσους διαχειρι... με τις σιδηροδρομικές εταιρείες. Επίσης, έκτο σημείο, διαχειριστές του δικτύου και ο ρόλο του ενισχύεται προκειμένου να υπάρχει σωστή αποτίμηση ε, των ε, επιδόσεών τους. Και έβδομο σημείο, οι ε, αρμοδιότητες του οργανισμού ρύθμισης, των ρυθμιστικών φορέων, έχουν ενισχυθεί επίσης. Όγδο σημείο και τελευταίο, η ανάπτυξη από την πλευρά της αγοράς κοινών συστημάτων ενημέρωσης και έκδοσης εισιτηρίων σωρευτικός, θα πρέπει να έχει χαρακτήρα προτεραιότητας προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη μετακίνηση των επιβατών με συνδυασμό διαφορετικών τρόπων μεταφορών και διασυνοριακώς. Ελπίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα υπάρξει συνένεση από πλευράς όλων για το αποτέλεσμα που επιτύχαμε από κοινού με μία προσέγγιση που από την πλευρά του Κοινοβουλίου ξεπέρασε και κάποιους πειρασμούς που θα ε, έφερναν δυσάρεστα αποτελέσματα για τι δικέ μα σιδηροδρομικέ εταιρείε. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει συνένεση και ελπίζω η δυνατότητα να εργαστούμε αποτελεσματικώ ε, ώστε να έχει ακόμα μεγαλύτερε δυνατότητε να είναι πραγματικά ευρωπαϊκό ο τομέα των σιδηροδρόμων όπω ελπίζει και η δική μα Επιτροπή να γίνει πραγματικότητα. Σα ευχαριστώ για τι συνεισφορέ σα. Danke sehr. Jetzt πολύ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να καταργήσουμε τον κανονισμό για τους λογαριασμούς των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποζημιωθούν αυτές οι εταιρείες για την πληρωμή υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει και που δεν χρειάζεται να καταβάλουν άλλα μέσα συγκοινωνιακά και μεταφορών. Για το θέμα λοιπόν αυτής της κατάργησης, εμείς θα προτείνουμε να ακολουθήσουμε τα όσα λέει η Κομισιόν, εκτός για τα όσα σχετίζονται με το τέταρτο παράρτημα, τέταρτη κατηγορία. Εκεί για τους λογαριασμούς, να σας πω πως οι κανονές θα πρέπει να ισχύουν και μέχρι τις 31 ε, Δεκεμβρίου του 2017, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν το χρόνο να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία για κάποια σχετικά κόστη, ε, για παράδειγμα για τις πεζοδιαβάσεις κτλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές, τη Γραμματεία, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάτι το οποίο κρίνω ε, ως μια εξαιρετική προσπάθεια συνεργασίας και αποτελεσματικότητας. Τώρα έχουν ζητήσει μερικοί το λόγο, αλλά επειδή έχουμε τέτοια τεράστια πίεση και έχουμε και το λεκτικό συνέδριο που πρέπει να μιλήσει και πριν από μισή ώρα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει, μόνο ένα λεπτό έκαστος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχει γίνει πολλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο από τα όσα μα προτείνει σήμερα ο κύριο Σασόν, για το σχέδιο σύσταση πάμε στη σελίδα 7 και θα δούμε ότι πολλέ φορέ μένει ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε αλλά πρέπει να σας πω εδώ έχουμε κάτι το οποίο θα έχει πολύ βαριές συνέπειες. Έχουμε μια δήλωση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου έχουμε σκοπό να κάνουμε μια επανερμηνία της συμφωνίας που είχαμε στον τριμερή διάλογο, το οποίο αποτελεί τριπλό λάθος για μένα. Καταρχήν, σε νομικό επίπεδο, σε τι αναφέρεστε στην δήλωση η οποία νομικά δεν είναι δεσμευτική και η οποία έχει ε, μπει στα εκτιμώντας. Αφήστε με να τελειώσω. Επιμένω λοιπόν το άρθρο 11. Μπορεί να μην είναι δεσμευτικό, αλλά έχει βαριές συνέπειες. Το άρθρο 11 λοιπόν, α, που λέει πώ έχουμε μια διάταξη που αντίκειται τελείως στο πνεύμα ολόκληρου του άρθρου 11. Δηλαδή, Έχουμε απόψει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή του Συμβουλίου που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεσμευτικά, ναι, αλλά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ξέρετε τι ειδικό βάρο μπορεί να έχει μια τέτοιου είδου δήλωση περί αντίστροφης θέση. Λοιπόν, τώρα, πριν ψηφίσουμε τον Ιούνιο ε, την α, ε, δήλωση του Τριμερούς και τη συμφωνία του Τριμερούς Δηλώους, σας δήλωσα εγώ ποια είναι η απόψή μου. Ε, και νομίζω ότι δεν μπορούμε σε τεχνικό επίπεδο να κάνουμε αυτό το σφάλμα. Και μετά υπάρχει και ένα ηθικό πρόβλημα, γιατί φανταστείτε να έκανε το ίδιο το Συμβούλιο. Θα φωνάζαμε πως πρόκειται για προδοσία. Γιατί είναι τελείως αντίθετο με την ε, συμφωνία, τη διοργανική που έχουμε μεταξύ αυτών των τριών θεσμικών οργάνων. Γι' αυτούς τους τρεις λόγους δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το κείμενο. Επρόκειτο να θέσω ακριβώς τα ίδια σημεία προς διευκρίνηση που έθεσε ο συνάδελφος μόλις τώρα. Η κυρία Ζάσκουν Ζάσκουν-Μπιλπάου. Μία ερώτηση έχω να κάνω για τον εισηγητή. Η έκθεση αυτή νομίζω αποτελεί το πρώτο σημείο το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό είναι η καινοτομία, γιατί όλα τα υπόλοιπα απορρέουν από αυτά που έχουμε στο πρώτο εδάφιο. Και επειδή έχουμε κάποια εμπειρία και ξέρουμε ότι εδώ και πολύ καιρό συζητάμε το πέμπτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους, να σας πω πως για τη διαλειτουργικότητα και επειδή ξέρουμε ποιες είναι αντιδράσεις των κρατών μελών και του Συμβουλίου και επειδή ξέρουμε ποια είναι η στάση του, σας ρωτώ το εξή. Όταν μιλάμε για άνοιγμα αγοράς, αυτές οι εξαιρεσει που αναφέρουμε, από ποιον θα αξιολογηθούν, από ποιον θα ελεγχθούν. Και αν η συμφωνία αυτή για το άνοιγμα της αγοράς μαζί με τις εξαιρέσεις ε, συμφωνηθεί, θα μείνουμε τελικά στην ίδια θέση που ήμασταν ή θα εφέρει κάτι διαφορετικό. Σας το λέω από περιέργεια. Γιατί θα ήθελα να γνωρίζω λίγο πιο πολύ τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή. Η κυρία ε, Τέλη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ διάβασα τις ε, συστάσεις του κυρίου Σασόλη και η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ σαφής. Όμως η έκθεση λέει να μην ξανανοίξουμε τη συζήτηση και να στηρίξουμε το κείμενο το οποίο προέκυψε από τον τριμερή διάλογο. Δηλαδή, η ομάδα μου που ήταν κατά στην πρώτη ανάγνωση, αν δεν αλλάξουμε τίποτα, δεν έχουμε κανένα λόγο να αλλάξουμε και θέση. Είναι τόσο απλό. Και θεωρώ πως είναι αρκετά παράξενο που ο κύριος ε, Σασόλη προτείνει μια αλλαγή με ένα παράρτημα για, την, ε, για το πλήρη άνοιγμα για τις υψηλές ταχύτητες. Με εκπλήσει αυτό και θα ήθελα να μου πείτε ουσιαστικά τι καθεστώς έχει αυτό το παράρτημα και επί της ουσίας δεν νομίζω ότι αυτή ακριβώς είναι και η ερμηνεία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε πολλά ερωτηματικά λοιπόν. Και θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Θα ξανανοίξουμε όλη τη συζήτηση, μόνο αυτό το κεφάλαιο. Για να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το κοινό που ταξιδεύει με τους σιδεροδρόμους. Ευχαριστούμε κυρία Αρνοτού. Ναι, ναι. Για την έκθεση, πρόεδρε, που σας είχα πει. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να επιταχύνω. Όπως ξέρετε και εγώ, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερως για το θέμα των δημοσίων κοινοφιλών υπηρεσιών, ιδίως των σιδηροδρόμων, που, ε, των οποίων άπτονται αυτές οι εκθέσεις για, το, για την ε, δέσμη των μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Εδώ βεβαίως βλέπουμε ότι εδώ ήταν λίγο σαν να έχουμε ένα μενού αλακάρτ για να ικανοποιηθούν όλοι, η αστική αριστερά, η δεξιά των επιχειρήσεων και οι ιδεολογίες της ακραίας αριστεράς. Αυτό όμως που με σοκάρει είναι ότι βλέποντας και το έργο της Επιτροπής υπάρχουν κυβερνήσεις που αντιτάχθηκαν και σε μέρη της οδηγίας που δεν είχαν να κάνουν με την πολιτική διάσταση, αλλά θα έπρεπε να έχουν τον χαρακτηρισμό του τεχνικού μέρους και θα μπορούσαν μάλιστα να χαρακτηριστούν και ως ε, ε, εξάρθρωση του σιδηροδρομικού κλάδου, έτσι όπως προτείνονται. Και επίσης Πρέπει να πω και το εξής. Εδώ παριστάνουμε ότι συμμετέχουμε στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, διευκολύνοντας τις διακρατικέ μεταφορές, αλλά καθόλου δεν κάνουμε αυτό λέγοντας προσπαθούμε να προκρίνουμε οικολογικές λύσει, προσπαθούμε να μείνουμε κοντά στη χώρα μας, να μην μετακινηθούμε πολύ. Αυτό θα ήταν πραγματική προσπάθεια για να μειωθούν οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Λέγεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται επιτρέπουν την πρόθεση των πραγματικών ε, ε, μεταφορών. Εγώ αυτό που διαπιστώνω στη Γαλλία είναι ότι υπάρχει κατάρρευση κατά 20% αυτών των εμπορευματικών μεταφορών τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν είμαι ευχαριστημένη και προσπαθώ να συμπυκνώσω αυτά που θα σας έλεγα, όμως προφανώς θα καταψηφίσω και τις τρεις εκθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε από την Επιτροπή ο κύριος Μπάλμπιν. Παρακαλώ σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το καταλαβαίνω απολύτω, Πρόεδρε. Θα είμαι άκρο συνοπτικό. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω όλη σα τη δουλειά για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, την τέταρτη δέσμη μέτρων για του Ε, Και πραγματικά φτάνουμε πολύ κοντά στο να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Εδώ θέλω να σταθώ σε μία πτυχή συγκεκριμένη και να διευκρινίσω μια δήλωση που έκανε η Επιτροπή προ το Συμβούλιο. Ε, κατανοώ τι ανησυχίε που εκφράστηκαν, αλλά πρέπει να τονίσω ότι εδώ μιλάμε για ένα σημαντικό πολιτικό συμβασμό στο Συμβούλιο. Μετά από απέτηση των 100 μελών να διευκρινιστεί πως εμείς και η Επιτροπή ερμηνεύουμε το ε, τα όσα δηλώθηκαν είναι ακριβώ το νομικό καθεστώ μια δήλωση. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Η δήλωση αυτή λέει ότι κατανοούμε ότι τα κράτη-μέλη ε, δύνανται να ε, θελήσουν βάσει των αρχών τη χρήση των γραμμών φυρμών υψηλή ταχύτητα το πώ θα τι χρησιμοποιήσουν, αλλά θα πρέπει οι ρυθμιστέ των σιδηροδρόμων να αποτιμήσουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ευχαριστώ και για τη συντομία. Και τώρα για να απαντήσετε θα δώσω σύντομα το λόγο στο Βίμ Βαντεγκάμπ και τους άλλους ηγητές. Ο Βίμ δεν θέλει, ο, ο κύριος Σασόλη. Ναι, εγώ θέλω. Πρώτα-πρώτα να τονίσω ότι καθόλου δεν θέλουμε να ξανανοίξει η συζήτηση που είχε να κάνει και με την θέση του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση. Σας καθησυχάζω κύριε Αντελή. Ως προς την παρατήρηση του κυρίου Μισελιέ και του κυρίου Άντερσον, της κυρίας Άντερσον, για το θέμα των υποχρεώσεων της Επιτροπής πρέπει να πω ότι όσοι παρακολούθησαν τον τριμερή διάλογο γνωρίζουν ότι το Συμβούλιο στο τέλος του τριμερούς διαλόγου προχώρησε σε δήλωση που ε, περιείχε την ε, δική του ερμηνεία για το άρθρο 11 κατόπιν αιτήματος ακριβώς του ίδιου του Συμβουλίου. Το άρθρο 11 αποτελεί μία λέξη specialis, ειδικό νόμο, ειδική διάταξη. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη διευκρίνησης εδώ. Είναι ε, συνηθισμένη πρακτική το Κοινοβούλιο να υποβάλει μετά την ψηφοφορία στο Στρασβούργο μια δική του δήλωση πάλι, η οποία ε, περιγράφει τη δική του ερμηνεία για το εν άρθρο. Εδώ μιλάμε για δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα ούτως ή άλλως, νομικός τουλάχιστον, και δεν μπορούμε μετά από 8 μήνε τριμερού διαλόγου να δεχτούμε μια δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητήθηκε από το Συμβούλιο, αλλά να μην αποκριθούμε με μια θέση του, του Κοινοβουλίου. Προσωπικώ, εγώ στο Κοινοβούλιο δουλεύω, εδώ βρίσκομαι, όχι στο Συμβούλιο. Όταν αλλάξω πόστο, θα ε, δεχτώ και αυτή τη δήλωση. Εμεί όμω ευαστήκαμε, καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία, Πρόεδρε, όσα μας ζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο και υπερασπιστήκαμε και το κύρος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο χρόνος. Σύντομα κύριε Άντερσον. Ε, ναι, το εκτιμώ αυτό που διευθυνέστηκε. Όμω, διαδικαστικά δεν περιελήφθηκε αυτό στα πρακτικά τη Επιτροπή τη 12 Ιουλίου όταν ψήφισε η Επιτροπή μα. Μήπω περιελήφθη, δεν ξέρω. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση, θέλω να πω Πρόεδρε, κυρία Μπιλμπάου, η διαδικασία είναι σαφή. Η προθεσμία για τι τροπολογίε 15 Νοεμβρίου στι 12 ε, το μεσημέρι. Θέλω να πω όμω ότι το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου τη Επιτροπή μα εγκρίθηκε ήδη στι 12 Ιουλίου. Έχει επιβεβαιωθεί. 12 Ιουλίου το ψηφίσαμε. Το Συμβούλιο στο μεταξύ ε, το επιβεβαίωσε επίσης σε πρώτη ανάγνωση. Οπότε οι τροπολογίες αυτές ουσιαστικά ε, και η προθεσμία είναι τυπικό ε, που πρέπει να το τηρήσουμε βέβαια αυτή τη διατύπωση. Βεβαίω μπορούν να κάνουν τα μέλη της Επιτροπής τροπολογίες για τη δεύτερη ανάγνωση, αλλά σε περίπτωση που εγκριθεί στο και μια τροπολογία ένα ο συμβιβασμό. Θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Οπότε, η διαδικασία αυτή είναι τυπική, θα γίνει, αλλά βεβαίως ο καθένας μπορεί να κάνει τροπολογίες, αλλά αυτή τη στιγμή εγκριθεί, πάει περίπατο όλος ο συμβιβασμός. Αυτό ήθελα να σας πω, γι' αυτό θέλω να σταματήσει εδώ η συζήτηση. Αυτές τι πληροφορίε χρειάζεστε. Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 15 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. φέτος. Εντάξει. Ε, Ευχαριστώ τους εισηγητές όλους για τη δουλειά που κάνανε προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου πάντα. Πρόεδρε, κυρία Μπελμπάο, συγγνώμη, έκανα μια ερώτηση εγώ στον κύριο Βαντεμκάμπ. Και δεν μου έχει απαντήσει κανείς. Θα ήθελα να μου απαντήσετε στη τόσο σαφή ερώτηση που σας έκανα. Και Ίσως μπορείτε να απαντήσετε γραπτά. Γιατί τέτοιου είδου θέματα πρέπει να διευκρινίζονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, δεν με πειράζει, μπορείτε να μου απαντήσετε γραπτά. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου μία απάντηση. Και γραπτά γίνεται, μπορεί μέχρι και διμερός να τα συζητήσετε. Αλλά είπαμε δεν θέλουμε γνωμοδοτήσεις. Αυτά που λέτε εσείς δεν με αφορούν. Λοιπόν,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 Please leave the room or sit down. Παρακαλώ ή βγείτε ή καθίστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση παρακαλώ σιωπή. Ακολουθεί η παρουσίαση τη ειδική έκθεση 816 του Ελεκτικού Συνεδρίου σχετικά με τι σιδηροδρομικέ εμπορευματικέ μεταφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπάλκο είναι ο κύριο ηγητή του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και ήρθατε και ιδιαίτερα που είχατε αυτή την υπομονή. Καθυστέρηση είχαμε με τις ψηφοφορίες μεγάλη, ήσασταν και παρόν εσύ στο τέλος. Ευχαριστώ για την κατανόηση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καλημέρα σας κύριε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της παρουσίασης της έκθεσης μου σε τριοδρομικές εμπορευματικές μεταφορές νομίζω ότι εντάσσεται στην ενδιαφέρουσα συζήτησή σας. Είναι χαρά μου που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου για τις τριοδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμη δεν βρίσκονται στο σωστή ε, ράγα. Ε, Ε, μετά την παρουσίασή μου στην Επιτροπή Κόντ 13 Ιουλίου, εκτίμησα την καλή συνεργασία που είχαμε με του συζητητέ κ. Μαρινέσκου και τα αξιόλογα σχόλια και συνεισφορέ από την κυρία Γιάλα Σέντερ και τον κύριο Λιμπεράτσκι. Ε, η σημερινή μου παρουσίαση ε, συνάδει με την ε, υπόσχεση του ελεγκτικού συνεδρίου να συνεργάζεται στενά μαζί σας με κάθε εξειδικευμένη κοινοβουλευτική επιτροπή για θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά μας. Σε αυτήν την έκθεση ελέγχου αποτεμήσαμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτελεσματικώς ενισχύσει τις αεροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Ε, πιο συγκεκριμένα είδαμε τις επιδόσεις αυτών των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχουν βελτιωθεί από το 2000 αποτιμήσαμε το στρατηγικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που έχουν σχεδιάσει η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και εξετάσαμε κατά πόσον τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στοχευθεί στις ε, κέρυες ανάγκες του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών όλα αυτά, ο συνεχιζόμενος έλεγχος για το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα Διαχείρισης ε, των Σιδηροδρομικών Μεταφορών πρόκειται να δημοσιευθεί το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά ήδη θα σας δώσω κάποια ε, εικόνα από τα βασικά της πορίσματα. Τώρα να στραφώ στην ειδική έκθεση 8-2016 για τι ιδεοδρομικέ και μεταφορές, μεταφορέ, ξεκινώντα με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμού. Οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από αυτέ τι μεταφορέ είναι 3,5 φορέ χαμηλότερε από κατά χαμηλέ ε, ω προ του τόνου ένα χιλιόμετρα από ότι οδικέ. Η προώθηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών είναι καθοριστική για την ε, πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι μεταφορέ εδώ και 25 χρόνια μεταξύ 2007 και 2013, ευρωπαϊκό προπολογισμό, συνεισέφερε 28 δισεκατομμύρια ευρώ στην χρηματοδότηση τέτοιων ε, προγραμμάτων. 75% τη ε, εσωτερική κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεχίζει να γίνεται μέσω οδικών μεταφορών. Το μερίδιο στην αγορά των εμπορευματικών κυκλοδρομικών μεταφορών να μειώθηκε από 19,7% το 2000 σε 17,8% το 2013. Κατά τη διάρκεια του ίδιου διαστήματος, το μερίδιο της χρήση συγκοινοδρομικών μεταφορών για εμπορεύματα στην Ελβετία αυξήθηκε κατά 40% ε, από το 2000 σε 48% το 2013 οι σιδηροδρομικές εμπορευματικέ μεταφορέ, ω βιώσιμη και φιλική ε, ως προς το περιβάλλον ε, μέθοδος μεταφοράς θα μπορούσε να μειώσει το κυκλοφορικό και το, τους, ε, τον αριθμό θανάτων που οφείλονται στι οδικές μεταφορέ. Το 2011 με τη Λευκή Βιβλία η Επιτροπή έθεσε ένα στόχο μετατόπισης 30% από τι οδικέ εμπορευματικέ μεταφορέ. ε, για αποστάσεις πάνω των 300 χιλιόμετρων, σε άλλους τρόπους ε, μεταφορών, όπως το σιδηρόδρομο ή τις πλωτές μεταφορές, μέχρι το 2030 και πάνω από 50% ε, μέχρι το 2050. Τι ε, διαπιστώσαμε λοιπόν. Συνολικά ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι επιδόσει των ε, σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν μη ικανοποιητικέ και το μερίδιο των οδικών μεταφορών έχει μεγαλώσει και άλλο από το 2000. Παρά του πολιτικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετατόπιση των εμπορευματικών μεταφορών από, από του δρόμου στο σιδηροδρομό, η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι υποδομέ δεν έδωσε τα αποτελέσματα που θέλαμε ε, και οι επιδόσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ τον όγκο και το μερίδιο αυτού του τρόπου μεταφορά δεν είναι αυτέ που στοχεύαμε. Μεταξύ 2000 και 2012 ε, ο όγκο των εμπορευματικών μεταφορών ετησίω παρέμεινε σχετικά σταθερό με 400 δι ε, τόνο χιλιόμετρων ενώ ο όγκος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αυξήθηκε από 1522 σε 1693 δις ε, τονοχιλιόμετρα. Έτσι, οι σιδηροδρομικέ εμπορευματικέ μεταφορέ τα τελευταία 15 χρόνια δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στι ανάγκε, ε, στον ανταγωνισμό μάλλον των οδικών μεταφορών, ενώ οι πλειοκτήτε ε, προτίμησαν τι οδικέ από τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Οι αρνητικέ αυτέ τάσει σε κάποια κατημέλη όπω την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία ευτυχώς ε, διαψεύστηκαν και εκεί αυξήθηκε η χρήση των σιδηροδρόμων. Παρά τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία 15 χρόνια για να βελτιώσει τι συνθήκε μεταφορά των αγαθών ε, με τον, ε, μέσω των σιδηροδρόμων, η απελευθέρωση τη αγορά έχει δημιουργήσει ανισότητα στην πρόοδο των κρατών και ένα ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο για την Ευρώπη ακόμη δεν φαίνεται κάπου στον ορίζοντα να δημιουργείται. Ε, το δίκτυο των σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ένα σύστημα κατακαιρματισμένων σιδηροδρομικών δικτύων που δεν ε, είναι διαλειτουργικά με πολλούς διαφορετικούς διαχειριστές υποδομών, ε, εθνικές αρχές ασφάλειας και ειδικού φορείς ρυθμιστικούς με διαφορετικούς κανόνες χρηματοδότησης, διαχείρισης, και τιμολόγησης κ.ο.κ. Επίσης, οι διάδρομοι για τις εμπορευματικές υδροδρομικές μεταφορές δεν προσαρμόζονται στις ανάγκες του κλάδου αυτού. Θα πρέπει να ε, υπάρξει καλύτερη ε, ανάμειξη των δύο τρόπων για τα εμπορεύματα και τους επιβάτες και να καλύπτονται και οι δύο κατηγορίες ε, σιδηροδρόμων και σειρμών. Οι οδικές ε, υποδομές είναι πιο εύκολα προσβάσιμες και δεν χρειάζεται να ε, πληρώνεται τέλος για κάθε χιλιόμετρο που διατρέχει ένας οδηγός. Ενώ αυτό ισχύει στους σιδηροδρόμους. Επιπλέον, η πρόσβαση στους σιδηροδρόμους με τα ανάλογα τέλη για τα εμπορεύματα είναι υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα, κέντρα, για τα τρένα, τα επιπληκτικά τρένα που συνδέουν για τα τρένα και τους προαστιακούς και μάλιστα περισσότερο από ότι η αντίστοιχη μεταφορά επιβατών. Οι τεχνικές και διοικητικές δυσκολίες ε, πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών με διαφορετικέ εθνικές διαδικασίες για την έγκριση του τροχαίου υλικού, τα πιστοποιητικά ασφάλειας, τις επιχειρήσεις ιδεοδρόμων, τις συλλογικές απαιτήσει για τους οδηγούς, για τα ζητήματα διαλειτουργικότητας, όλα αυτά τα οποία ε, φροντίζουμε, ε, θα φροντίσουμε να ε, επισημάνουμε στην επερχόμενη έκθεσή μας. Ε, Όπω σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τρία ή πέντε κράτη-μέλη τα οποία επισκεφθήκαμε στι αποστολέ ελέγχου για να δούμε τι έχει διατεθεί στις οδικές μεταφορές και τις συνδρομικές από το 2007 μέχρι το 2013 μέσω των ε, ταμείων συνοχής ε, είδαμε εκεί ότι τελικά δεν στοχεύτηκαν συγκεκριμένε συνδρομικέ εμπορευματικές ανάγκες αλλά περισσότερα οι ανάγκες ανάμειξης ή μεταφοράς επιβατών. Τέλο, η κακή συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου επηρεάζει τη βιωσιμότητα και τι επιδόσεις των υποδομών που ε, ε, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σειρμοί που πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τρένα εμπορευματικών μεταφορών, αλλά με περισσότερες δυσκολίες και περιορισμούς στην ταχύτητα σε σχέση με τα επιβατικά. Αυτό επηρεάζει και το δίκτυο συνολικά, αλλά και τον όγκο των αγαθών που μεταφέρονται. Κυρίε και κύριοι, βασιζόμενοι στα άνοθη πορίσματα. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρξε αποτελεσματική στο να ενισχύσει τι δεδομικέ εμπορευματικέ μεταφορέ. Απέτυχε τα τελευταία 15 χρόνια να βρει μια επαρκή απόκριση στι ανάγκε ανταγωνισμού των οδικών μεταφορών. Οι μεταφορέ εμπορευμάτων στου σιδηροδρόμου, παραμένουν μη ικανοποιητικέ ως προς την ανάμειξη διαφορετικών τρόπων, τους όγκους και τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν, ακόμη και αν κάποια κράτη-μέλη βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Τα στρατηγικά και ρυθμιστικά ζητήματα που συντοπίζονται στην εκθεσή μα δεν καλύφθηκαν ούτε με επιπλέον χρηματοδότηση και αυτή έτσι κι αλλιώ μόνη τη δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Βάσει αυτών των συμπερασμάτων, το συνέδριο προτείνει στην Επιτροπή και τα κάτι μέλη να ακολουθήσουν τι ε, ε, εξή δράσει προκειμένου να βελτιώσουν το στρατηγικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ε, εντό του οποίου γίνεται η μεταφορά αγαθών μέσω σιδηροδρόμων και να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σύσταση πρώτη. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί ρυθμιστέ διαθέτουν και μπορούν πραγματικά να ασκήσουν τι απαραίτητε αρμοδιότητε με ανεξαρτησία και του απαραίτητου πόρου, ιδιαίτερω για να αντιμετωπίσουν τι πρακτικέ που πλήττουν τον ανταγωνισμό. Σύσταση 2. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν του κανόνε διαχείριση τη ε, κυκλοφορία, τι ειδικέ ανάγκε του τομέα εμπορευματικών μεταφορών, λόγω χάρη ό,τι αφορά τα ε, χρονοδιαγράμματα, τη διάθεση ε, ε και σύρμων και την ποιότητα αυτών. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών σε όλη την Ευρώπη για του διαδρόμου εμπορευματικών μεταφορών. Ε, σύσταση 3. Η Επιτροπή μαζί με τα κατημέλη θα πρέπει να απλουστεύσουν και να εναρμονίσουν τι διαδικασίε για την έκδοση τροχαίου υλικού και για την έκδοση πιστοποιητικών ασφάλεια για τι επιχειρήσει ιδιοδρόμων. Η έκθεσή μα αναφέρει ξεκάθαρα την ανάγκη σύντομη έγκριση του τέταρτου πακέτου για του υδροδρόμου και με μεγάλη ικανοποίηση γιατί στον μεταξύ αυτό έχει γίνει πραγματικότητα ε, σε ό,τι αφορά τον τεχνικό πυλώνα του πακέτου ε, και ελπίζω ότι και ο πυλώνας της αγοράς θα φτάσει ε, τον Ιούλιο στην Επιτροπή, που έφτασε στην Επιτροπή σας τον Ιούλιο, θα ψηφιστεί σύντομα. Ε, θα γίνει αμελητή ελπίζω αυτό και βάσει τη σύσταση 3 η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να αποτιμήσουν την ε, δυνατότητα να προχωρήσουμε στην απλούστευση των γλωσσικών απαιτήσεων για τους οδηγούς ε, σιδηροτροχιών. Ε, η Σύσταση 4. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί ε, συστηματικά την πρόοδο προς τους στόχους που εντόπιζε η Λευκή Βιβλία στο 2011 για τη μετατόπιση των μεταφορών από τους δρόμους προς τους σιδηροδρόμους για τη μεταφορά αγαθών με συγκεκριμένα έγγραφα και έντυπα που καθορίζουν την πολιτική μας. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να ικανοποιούν τις ανάγκες όσων μεταφέρουν εμπορεύματα είτε είναι επιλεκτήτες είτε άλλοι χρήστες για να υπάρχουν καλύτερες, καλύτερες ποιότητες υπηρεσίες. Σύσταση 5. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ένα σύστημα ίσων κανόνων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορών μεθόδων ε, μεταφορών με επιπλέον ρυθμιστικέ διατάξει, προκειμένου να προωθηθούν οι πραγματικέ μεταφορέ μέσω σιδηροδρόμων. Σύσταση 6. Η Επιτροπή και τα κάτι θα πρέπει να προβλέψουν την απαραίτητη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ε, για, την, για τις υποδομές των μεταφορών ε, προκειμένου να συνάδουν οι στόχοι αυτοί με τους πολιτικούς στόχους με ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών για τα εμπορεύματα και αντιμετωπίζοντας τα συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν κυκλοφορικέ δυσκολίε, αλλά και να βελτιωθούν και συνδέσει των σιδηροδρόμων με λιμένε και σε διασυνοριακέ περιοχέ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί κατά πόσο η χρηματοδότηση αξιοποιείται σωστά σε προγράμματα ε, επενδύσεων για τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Σύσταση 7. Τα κάτι μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσουν τον συντονισμό των ε, σιδηροδρομικών επενδύσεων προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και να αποφύγουν την ανάπτυξη του ε, δικτύου με τρόπο κατακαιρματισμένο. Θα πρέπει να αξιοποιήσουν την δυνατότητα κάθε έργου να αυξήσει συνολικά τι επιδόσει του ε, συστήματο μεταφορά εμπορευμάτων με συστηματική συμπερίληψη ποσοτικών στόχων για αυτέ τι μεταφορέ προκειμένου τα έργα να υλοποιηθούν σωστά. Σύσταση 8 τελευταία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, να βεβαιωθούν για την σωστή συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, ιδίω ό,τι αφορά του διαδρόμου εμπορευματικών μεταφορών. Η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, και προστατεύουν με συστέ στρατηγικέ ανάπτυξη αυτά τα δίκτυα και τι υποδομέ του. Κύριε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και πραγματικά αναμένω με υπομονησία τα σχόλια και τι ερωτήσει σα. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την υπομονή που δείξατε, για την παρουσίαση και την ανάλυση σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε μερικούς βουλευτές που ενδιαφέρονται και σίγουρα έχουν και σχόλια όσο και ερωτήσεις να σας κάνουν. Πρώτος, ο Βιμ Βανενκάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και τον κύριο Μπάλκο και το επιτελείο του ε, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οφείλω να ομολογήσω ότι δυστυχώς, δυστυχώς η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που ξέραμε κι εμείς και μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, τα διαπιστώνουμε. Ωραία λέει, τα λέει η πολιτική για την αλλαγή ε, των μεταφορών, δηλαδή για ε, να βοηθηθούν και άλλα μέσα μεταφοράς από τον αυτοκινητόδρομο. Αλλά ο αυτοκινητόδρομος κυριαρχεί θα πρέπει να επανέλθει στο σωστό του μέγεθος, στις σωστές του διαστάσεις, γιατί έχει διωγγωθεί υπέρμετρα ο κλάδος των οδικών μεταφόρων. Έχω μερικές παρατηρήσεις. Πρώτον, κύριε Μπάλκο, μπορείτε να μας πείτε κάτι για τα δικαιώματα των καταναλωτών. των Χριστών μάλλον και βλέπουμε ότι αυξάνονται τα τέλη ε, για διάφορους λόγους και αυτό δεν βοηθάει τις εμπορευματικές μεταφορές. Δεύτερον, κοιτάξτε τίποτα για την ψηφιοποίηση, γιατί εμείς ξέρετε στον κλάδο των μεταφορών ε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη ψηφιοποίηση. Αυτό βοηθάει τις εμπορευματικές μεταφορές ή όχι. Και τρίτη ερώτηση, COP21, ε, Συμφωνία για το κλίμα. Όλο και περισσότερο ε, μας βάζουν ε, διάφορες υποχρεώσεις για να γίνουν πιο βιώσιμες οι μεταφορές σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Αυτό το έχετε μελετήσει στην έκθεσή σας. Ε, μετά, διασυνοριακά προβλήματα, τα γνωρίζουμε και αυτά. Εκπλήσωμε που στους διαδρόμους των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ε, οι υποδομές και πάλι επιμένουν πάρα πολύ στον αυτοκινητόδρομο και όχι στο σιδηρόδρομο. Μήπως να το συζητούσατε αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επανέλθει ε, αυτό ε, το θέμα της ισορροπίας. Και ρωτάω κάτι και για το θόρυβο τώρα, για την ηχορύπανση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ε, συνδρομικές μεταφορές είναι ο θόρυβος μπορούμε να το ξεπεράσουμε για να ε, προωθηθεί αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ για τις 8 συστάσεις, αλλά μία είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Για μας είναι πρόβλημα. Ε, εγώ κυκλοφορώ πολύ με το τρένο και δεν θέλω να είναι ε, ε, η προτεραιότητα πρώτα τα εμπορεύματα και μετά οι ε, επιβάτες. Πρώτα οι επιβάτες και μετά τα κοντέινερ. Ευχαριστώ η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το συνάδελφο του Ελληνικού Συνέδριου για την παρουσίαση που έκανε και να ευχαριστήσω και την ομάδα του. Έχω την αίσθηση ότι τα έχουμε ξαναπεί όλα αυτά και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και πάλι επαναλαμβάνει αυτό που μας έχει πει στο παρελθόν. Οι εκθέσεις λοιπόν που έχουμε προετοιμάσει για να αντιμετωπίσουμε το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο και κυρίως το τεχνικό σκέλος, όπου και ο πρόεδρος και εγώ ήμασταν εισηγητές και για τη διελειτουργικότητα και για την ασφάλεια σε διαφορετικές γνωμοδοτήσεις, πάντοτε σκοντάφτουν σε θέματα τα οποία μόλις εξηγήσετε εσείς τώρα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τα κράτη-μέλη. Γιατί ακόμα και το 2013 που κάναμε την αναθεώρηση των ε, κατά priority ευρωπαϊκών κατά προτεραιότητα ευρωπαϊκών ε, έργων όπου μιλήσαμε για συμφόρηση ε, για το γεγονός ότι οι οδικές μεταφορές έχουν ε, φτάσει σε ωριακές καταστάσεις. Είδαμε ότι δεν υπήρξε καθόλου ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη. Εξακολουθούν να έχουμε τα σύνορα κλειστά, εξακολουθούμε να έχουμε αυτές τις ωριακές καταστάσεις και πάλι δεν έχουμε χρηματοδότηση. Γιατί δίνεται προτεραιότητα από όλα τα κράτη-μέλη σε άλλα θέματα. Και θα ήθελα κάποιο να μου απαντήσει, αν μπορεί κάποιο, τι να κάνουμε πια. Νομίζω ότι έχουμε βαρεθεί. Τα έγγραφα, τις εκθέσεις, τα στοιχεία, όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται γύρω μας. Τι μπορούμε να κάνουμε πια. Και εντωμεταξύ γινόμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί, δεν κάνουμε αρκετές καινοτομίες, τα φορτηγά εξακολουθούν να ρηπαίνουν στο δρόμο και παράλληλα εμείς συνεχίζουμε να εγκρίνουμε εκθέσεις για να μειώσουμε τις εκπομπές και ζητάμε από τις εταιρείε που είναι βιομηχανικές, οι οποίες μπορούν να μας βγάλουν από αυτή την κατάσταση, να κάνουμε μια προσπάθεια και τις τιμωρούμε όλο και παραπάνω με τα δικαίωμα εκπομπών. Σε ποια δημοκρασία πήγαν, πόσα αγόρασαν, πόσα πούλησαν και τι θα γίνει για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουν οι οδικέ μεταφορέ να αυξάνουν του ρήπου που εκλείνουν στην ατμόσφαιρα. Μιλάμε για μια μεγάλη αντίφαση. Σίγουρα δεν χαίρεστε που με ακούτε, αλλά επιτρέψτε μου να σα ρωτήσω και πάλι τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν αρκετέ χώρε οι οποίε στοιχημάτισαν υπέρ των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και εκεί είναι καλύτερα τα αριθμητικά στοιχεία και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν τα κράτη στα οποία αναφερθήκατε εσείς βελτίωσαν τον, τις εσωτερικές μεταφορές ή ανέκαναν και προσπάθειες για τις διασυνοριακές μεταφορές και μιλώ πάντα για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Δηλαδή αυτή η βελτίωση στην οποία αναφερθήκατε είναι μέσα στη χώρα τους ή σε σχέση με τις υπόλοιπε χώρες με τις οποίες έχουν αυτή τη διασυνοριακή σχέση γιατί η λεπτομέρεια αυτή είναι πολύ σημαντική και γιατί έτσι θα έχουμε και κάποιες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει εμείς στα ευρωπαϊκά οργάνα προσπαθούμε να προχωρήσουμε προ μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ανταποκρίνεται στι απαιτήσει των κλάδων όλων των κρατών μελών και παράλληλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν και μιλώ για τις κυβερνήσεις τους, τις των 28 που προσπαθούν να βρουν μηχανισμούς για να προστατεύσουν και πάλι και να γίνουν πιο κερδοφόρες οι ίδιες τους οι μικρές αγορές η εμπειρία μου με οδηγεί στο να ρωτώ τι πια μπορούμε να κάνουμε. Εκτός από τις συστάσεις δηλαδή τις δικές σας, θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα διαχειριστείτε εσείς αυτές τις συστάσεις. Θα διαπραγματευτείτε με τα κράτη-μέλη, θα κάνετε κάτι αντίστοιχο, μπορούμε να σκεφτούμε κάτι. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός για να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνω σε τι χρησιμεύουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές όχι γιατί δεν προσπαθούμε εμείς, αλλά γιατί δεν μας ε, ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Τι θα κάνετε εσείς με τις συστάσεις σας, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Έχω βάλει και το δικό μου όνομα στη λίστα και μετά μπορείτε να απαντήσετε. Νομίζω πολιτική βούληση υπάρχει, αλλά προς τη λάθος κατεύθυνση. Εδώ και χρόνια και δεκαετίες έχει μαγιάσει η γλώσσα μας στο Κοινοβούλιο ε, όλες οι πολιτικές ομάδες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα. Εσείς μας επιβεβαιώνετε στις εκθέσεις σας για τις εμπορευματικέ μεταφορές, στο σιδηρόδρομο ή και στις οδικές μεταφορές και όλα αυτά και τα διασυνοριακά. Αλλά στην Ευρώπη έχουμε κάποιες προϋποθέσεις και ένα πλαίσιο που η ε, πολιτική βούληση λέει δρόμος, δρόμος, δρόμος, αυτοκινητόδρομος και φουλ αυτοκινητόδρομος και κάθε μέρα ε, και ε, που περνάει ε, αυξάνεται ο αθέμητος ανταγωνισμός εις βάρος του σιδηροδρόμου και ευνοώντας τους αυτοκινητοδρόμους. Κάνατε αναλύσει για τα χρήματα από τα διορθωτικά ταμεία. 60% πάει στον αυτοκινητόδρομο, 20% στο σιδηρόδρομο. Εμεί στο Κοινοβούλιο είχαμε πλειοψηφία που έλεγε τουλάχιστον το 40% να πηγαίνει στο σιδηρόδρομο. Τα στείλωσε το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως όταν έχει δυνατότητες επιλέγει τον αυτοκινητόδρομο. Το ταμείο ΕΦΣΥ 75% πάει στο αυτοκινητόδρομο. Τρία ήταν τα έργα για τα τρένα. Από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αυξάνεται ο ανταγωνισμός και στραγγαλίζεται ο σιδηρόδρομος. Και έχουμε και τα διόδια. Αναφέρεται την Ελβετία. Η Ελβετία έχει τα πιο ψηλά διόδια, τριπλάσια από τη Γερμανία για τον αυτοκινητόδρομο και τα λεφτά τα παίρνουν και τα δίνουν στο τρένο. Γι' αυτό έχουν 100% ε, ηλεκτρικά τρένα περίπου. Στη Γερμανία συγκριτικά είναι 60%. Παρόλο που αποφασίστηκε εδώ και 100 χρόνια και πλέον στη Γερμανία να ε, έχουμε ηλεκτρικά τρένα. Τίποτα δεν γίνεται. Στα διασυνοριακά τα ίδια. Είπατε θα μπορούσαμε από το σύνορο μέχρι τον επόμενο κόμβο να πάρουμε ενίσχυση μέχρι το 85% από τα διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία συνοχή. Δεν τα κάνει η Κομισιόν αυτά. Αυτό είναι αποφασιστικό όμω για τι χώρε. Οι χώρε είναι σωστρεφείς, γιατί κοιτάνε τα εθνικά του σύνορα από τα σύνορα προ τα μέσα, όχι προ τα έξω. Εμεί όμω μιλάμε για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και η Κομισιόν αυτά θα πρέπει να κάνει. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ακόμα και ο Γερμανός υπουργό Μεταφορών μπορεί να έλεγε δεν με νοιάζει να βελτιώσω τις συνδέσεις με την ε, Γαλλία, την Ολλανδία και την Πολωνία, αλλά αν μου δώσετε ευρωπαϊκά λεφτά θα το κάνω. Αθέμητος ανταγωνισμός, επαναλαμβάνω, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη αποφάσισαν κάθε μηχανή σύρμου να πληρώνει ε, ένα είδος τέλους, ένα είδος ε, διοδίου για κάθε χιλιόμετρο. Στον αυτοκινητόδρομο αυτό εναπόκειται στα κράτη-μέλη και επιβάλλουν 1% ε, του δικτύου, στο 1% του δικτύου διόδια, ενώ στα τρένα 100%. Ωραία τα κηρύγματα της Κυριακής από τα μπαλκόνια. Στην πράξη τι κάνουμε, εσείς πώς θα επηρεάσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αντιδράσει. Γιατί και εμείς προβληματιζόμαστε και ο κύριος Ρόιτερς θα πάρει μέσα το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός τα ξέρει και μπορεί να σας τα πει. Έχουμε ευθύνη όλοι. Εμείς πιέζουμε για τα διασυνοριακά έργα και θα πρέπει να το κάνουμε, διότι δεν πρόκειται να πετύχουμε κανένα κλιματικό στόχο αν το 75% των εμπορευμάτων και παραπάνω συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους. Στην Ευρώπη νομίζω έχουμε 17% εμπορευματικές ή δρομικές μεταφορές ενώ 40% οι Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι και η κατεξοχήν χώρα που βασιλεύει το αυτοκίνητο και μας βάζει τα γυαλιά η Αμερική. Ε, χειρότερη ξεφτύλα δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ για την Ευρώπη. Ο κύριος Ρόιτερς τώρα, τον Παλάκη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να γνωμοδοτήσει, γνωριζόμαστε. Αλλά για να δούμε τώρα πώς μπορείτε να βοηθήσετε το ελεκτικό συνέδριο έτσι ώστε να είναι καλύτερη η έκθεσή του του χρόνου. Έχετε το λόγο. Yeah. Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί εκπρόσωποι του Ελληνικού Συνεδρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που έχω το λόγο και μπορώ να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί γενικότερα με το Ελληνικό Συνέδριο για το τι θα συμβεί ε, στο μέλλον ε, για τη σιδηροδρομική αγορά στην Ευρώπη που ακόμα είναι σε μη ικανοποιητικό επίπεδο. Βεβαίως, ε, ε, θα απαντήσουμε στις συστάσεις σας και πρέπει να σας πω πως η σύσταση, οι συστάσεις αυτές φτάνουν την κατάλληλη στιγμή γιατί στηρίζουν προφανέστατα τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναζωπυρώσουμε το σιδηροδρομικό κλάδο και έχουμε μια σειρά από μέτρα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν εξελίξη. Τα γνωρίζετε κι εσείς πως Αξιολογούμε τον κανονισμό για να δούμε αν και ο κώδικας λειτουργίας και το κανονιστικό πλαίσιο χρειάζονται βελτιώσεις και επίσης παρακολουθούμε και τη διαδικασία της δήλωσης του Ρότερνταμ για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη πρόοδο τώρα και να μην περιμένουμε τη στιγμή της αναθεώρησης που θα γίνει ε, του κανονισμού για τις εμπορευματομεταφορές μέσω σιδεροδρόμων στο μέλλον. Επίσης, ακούστηκαν κάποια σχόλια από την κυρία Πιλπάκη και από εσάς κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να τονίσω πως έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, ακόμα και σήμερα το πρωί εδώ, για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο με τους τεχνικούς και πολιτικούς πυλώνες, τον πυλώνα της αγοράς, δηλαδή τα σκέλη αυτά, τα οποία ελπίζουμε πως θα οδηγήσουν σε αυτά αποτελέσματα. Ελπίζω πως όλες αυτές οι κοινέ προσπάθειες θα μας δώσουν ε, πιο ισχυρές εμπορευματομεταφορές ε, σιδηροδρομικές στο μέλλον. Θα ήθελα να απαντήσω στα όσα είπαν ο συνάδελφος κ. Βανδεκάμ και εσείς για το κατά πόσο πως υπάρχει ε, ε, πολύ μεγάλη επένδυση από το Connecting Europe ε, στις, ε, στις οδικές μεταφορές. Νομίζω ότι σε αυτό λαθεύεται. Είναι γύρω στο 4% Όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν για περιβαλλοντικά ε, φιλικά μέσα συγκοινωνία, όπω για παράδειγμα έξυπνα δίκτυα, πλωτέ μεταφορέ, σιδηροδρομικέ συγκοινωνίε και μεταφορέ. Και να σα πω επίση πω και στα πλαίσια της συνοχής κάνουμε κάτι αντίστοιχο και η χρηματοδότηση η οποία που είναι διαθέσιμη είναι πάντα 50-50 με κατανομή τέτοια ανάμεσα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Θα θέλαμε να είναι παραπάνω. Τώρα για τα διασυνοριακά ε, Έχουμε μιλήσει για ποσοστά συγχρηματοδότηση όταν μιλήσαμε για τον κανονισμό για το Connecting Europe Facility που είχαμε ε, για τις χώρες συνοχής 85, για τους υπόλοιπους 80-40 λέει ο μιλητής. Και είχαμε πει να πάμε στο 85 έτσι ώστε κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη βούληση να πράξουν κάτι αντίστοιχο και να μπορούν και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να, να ε, εφαρμόζουν αυτά τα διασυνοριακά έργα. Βεβαίως το πώς μπορούμε να έχουμε ένα πιο δυναμικό κλάδο στις σιδηροδρομικές συμπορομεταφορές στην Ευρώπη είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Έχουμε κατά θέση και το πακέτο και τον κανονισμό και σίγουρα στη θέση του κ. Μπάλκο και τις ομάδες του ε, την κατάλληλη στιγμή ήρθαν έτσι ώστε να παραδώσουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα. Ευχαριστώ. Τώρα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε στις ερωτήσεις και τα σχόλια της Επιτροπής. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχετε κάθε δίκιο. Και κύριε Μπιλπάου και κύριε Βαντερκάμ, έχετε απόλυτο δίκιο και εσείς κύριε Πρόεδρε. Είστε ευρωβουλευτές και είναι πολύ σημαντικά τα καθηκοντά σας σε νομοθετικό επίπεδο και θίξατε κάποια θέματα σχετικά καταρχήν με ε, τα τέλη πρόσβασης, με την ψηφιοποίηση, ε, με τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε ε, διασυνοριακά. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συνεργασία με αυτήν είναι ένα θέμα που σας απασχόλησε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την ευκαιρία να λάβει η θέση κατά την, κατά την παράθεση διαδικασία και να σας πω πως ε, στους ελέγχους που κάναμε για την απόδοση ε, λάβαμε υπόψη και τις ε, απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία συμφώνησε με κάθε μία από τις συστάσεις μας. Οκτώ συστάσεις και συμφώνησε για όλες. Άρα ευθυγραμμίζονται οι απόψεις μας και τι θα έπρεπε λοιπόν να πράξουμε παραπάνω. Εμείς κάνουμε αυτούς τους ε, ελέγχους απόδοσης που αποτελούν ε, τμήμα της ετήσιας έκθεσης που αποτελεί ένα εργαλείο για τη διαδικασία απαλλαγής. Και αυτό συνδέει τις προσπάθειες που κάνει και ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε εμείς στέλνουμε αυτή την έκθεση Και θα χαιρόμουν πολύ αν κάποιο μέλος ε, της ε, ομάδας μου θα μπορούσε να απαντήσει και τις πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Ο Ούρμπανης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να συμπληρώσω τα όσα είπε ο κύριο Μπάλκο για τα τέλη πρόσβαση και για το θέμα του κύριου Βαντενκάμ. Να σας πω πως παράγραφος 68 με 73 της έκθεσης αναφέρεται σχετικά και κυρίως παράγραφος 73 όπου δίνουμε όχι μόνο το παράδειγμα της ε, Ελβετίας αλλά και της Αυστρίας. Και αναφέρουμε πω. και άλλες μέθοδοι που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις ιδεροδρομικέ εμπορευματομεταφορές. Τελευταία μου παρατήρηση για το τι μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, οι συστάσεις θα κατατεθούν και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και παρακολουθούμε και την ε, εφαρμογή της σύσταση και αυτό το κάνουμε σε κύκλους 2-3 ετών. έτσι ώστε όλες να ε, τύχουν τις κατάλληλες παρακολούθησης και να εφαρμοστούν όπως πρέπει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε και αυτό το θέμα στη μέσα διάταξη. Βλέπουμε ότι έχουμε κοινή θέση. Ε, το θέμα είναι τι να κάνουμε. Ωραία τα λόγια. Αλλά θέλουμε να δούμε και έργα. Δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από δεκαετή και μεγαλύτερη πίεση κάπως κουνήθηκε σε ό,τι αφορά ε, ε, τα θέματα αυτά. Θετικό είναι. Ε, καλή επικοινωνία έχουμε. Για να δούμε τώρα θα βγει και τίποτα. Είναι καλύτερη επόμενη έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθατε και περιμένατε τόση ώρα. Αλλά Είχαμε μια συζήτηση για το πακέτο αυτό το συνδρομικό. Ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Κάνε μια μικρή υπέρβαση ωραρίου. Πάμε στα διάφορα που δεν έχουμε. Επόμενη συνεδρίαση 5η Δεκεμβρίου, μέρα Δευτέρα, ε, στις 3 ε, το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.